Dear colleagues, we will start with the committee. Please sit. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Comenzamos con la, con la reunión de, de esta mañana. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρωινή μας συνεδρίαση. Παρακαλώ, Ξεκινάμε λοιπόν με την πρωινή συνεδρίαση. Καταρχάς να σας πω ότι υπάρχει μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Εχθές το απόγευμα δεν μπόρεσε να συζητηθεί το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης ε, του πολιετούς δημοσιονομικού πλησίου 2014-2020, διότι η συντάκτρια της γνωμοδότησης δεν ήταν εδώ. Επομένως, ε, η συζήτηση θα είναι το τελευταίο σημείο που θα συζητηθεί στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Επίσης, στον κατάλογο ψηφοφοριών συμπεριλαμβάνουμε και την ε, ε τροπολογία για το gender mainstreaming του μηχανισμού. Αυτού δεν το είχαμε, θα το συμπεριλάβουμε και αυτό στις ψηφοφορίες. Εντάξει, ξεκινάμε λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Έχετε όλοι τις κάρτες ψηφοφορίας. Eh, Ξεκινάμε με την εφαρμογή της οδηγίας 2011 της 5ης Απριλίου του 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων με γνώμονα την ισότητα των, φόλων, ε, των φύλων. Τροπολογία 88. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 8. Υπέρ, καταπίπτει, συγγνώμη, καταπίπτει. Τροπολογία 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε μια επαλήθευση της 94. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η 49 θα ψηφιστεί ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, δεν καταλαβαίνω. Να κάνουμε μια επαλήθευση για την 99. Πώς Είναι ε, ήταν προφανέστατο. Εγώ μάλλον δεν είδα καλά σε αυτή την περίπτωση. Εγκρίνεται. 5 ε, της ΛΥΜΠΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε στην 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται θα ήθελα να σας ζητήσω να σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν σήκωσε κανείς σε αυτή την περίπτωση. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα. Ε, es que ahí ya no llego. Ε, μέχρι εκεί δεν μπορώ να το βρω. Κατα... Απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ο κύριος ε, Ταραμπέλε θέλει επαλήθευση του τρίτου τμήματος. Ωραία. Επαλήθευση για το τρίτο τμήμα. Ε, ορίστε, κύριε Ταραμπέλα, εγώ βλέπω καλύτερα από εσά. Εγκρίνεται. Μικρόφωνο, πρόεδρος. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε. Αφού δεν σηκώνετε τα χέρια σας θα επαληθεύουμε. 108. 108. Εγκρίνεται. Η 48 της Λιμπέ καταπίπτει 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε μια επαλήθευση της 109. 109. Απροβάδα. Εγκρίνεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 22, δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές να επαληθεύσουμε την 130 Έρχεται η ψηφοφορία. Se cierra. Rechazada. Απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 133 αποσύρθηκε. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε την 135. Άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιος δεν ε, ψήφισε. Έχετε την κάρτα σας, δεν έχετε ψηφίσει. Εγκρίνεται. 136. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 149 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 160 αποσύρθηκε, 161 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 169 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 170 κατά καταπίπτει, συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, Περνάμε στη λίμπα 39, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 171 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 172 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 100, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, να το επαληθεύσουμε, το δεύτερο τμήμα της 172, άρχεται η ψηφοφορία. Ρετσαφάδα. 170... Απορρίπτεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ε απορρίπτεται. 176 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θα ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 176. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα. Συμβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 181 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές ε, έχω αποπροσανατολιστεί τελείως σήμερα να κάνουμε μια επαλήθευση 183 άρχεται η ψηφοφορία Se cierra Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Είναι σε κάποιες περιπτώσεις πολύ κοντά οι διαφορές και είναι δύσκολο να το δω με το μάτι. 186. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 180... 85 επαλήθευση. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε μια επαλήθευση για την 188. Εγκρίνεται. Λίμπε 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 195 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, το δεύτερο τμήμα καταπίπτει, συγγνώμη, γιατί εγκρίθηκε το, το 194. Παράγραφος 30, καταπίπτει και αυτό, 196 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται, συγγνώμη, 197 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 198 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, λίμπε 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 203 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 202 υπέρ. Καταπίπτει. Όχι, δεν καταπίπτει γιατί απορρίφθηκε. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 200 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λίμπε 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 205 καταπίπτει, 206 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 207 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λίμπε 33 υπέρ, Κατά. Επαλήθευση για τη 207. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 208 καταπίπτει. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας. Διότι βλέπω πολύ καλύτερα. Θα σας βάζω κάποιον να κάθετε εδώ για να βλέπετε τι τραβάω. Συμβαστική τροπολογία 16 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε μια επαλήθευση. Sí. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 215 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 229 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 19 δεν ψηφίζεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ.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 234 υπέρ, κατά, αποχές εκρίνεται. 235 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές, δεν ε, βλέπω να το επαληθεύσουμε. Γιατί 237, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Λίμπε 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 47 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 241 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λίμπε 44 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε σε αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται ή 5 κατά πι. Την 5 ως προσθήκη, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά, αποχές, επαλήθευση για την εννέα. Σε cierra Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. δέκα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. έντεκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 18 αποσύρθηκε, συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 23 υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, λίμπε 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω. Γιατί οι περισσότεροι νομίζω απήχαν. Ψηφίζουμε την 57. Απροβάδα. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η ε, αιτιολογική σκέψη B της ΛΥΜΠΕ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F υπέρ κατά αποχές, εγκρίνεται. G υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Λίμπε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Pues aprobado por 26. Εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ, καμία κατά και 6 αποχές. Συγχαρητήρια, κυρία Μπίρτερ. Madre mía, hoy tenemos votos gorditos, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, que tenemos una mañana interesante. Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρον πρωινό ψηφοφοριών. Κουράγιο όλοι και να ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Αρένα. Φτώχεια μια προοπτική με γνώμονα το φύλλο. Ξεκινάμε λοιπόν. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε για την 107. Κατά Καταπίπτει. Λυπάμαι κύριε Σεμπαστιά. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλε 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εκατόν δεκαεννέα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να κάνουμε μια επαλήθευση για τη συμβαστική τροπολογία 2. Ναι, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 145 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Για το πρώτο τμήμα της 145. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146, 147 και 148 που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρω, για να κάνουμε μια επαλήθευση. 146, 147, 148. Απορρίπτονται. 149 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 163 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 173 υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε την 173, άρχεται η ψηφοφορία. Απροβάδα. Εγκρίνεται. 174 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλεφτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 179 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 180 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 181 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 184 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έμπλη 13 α, συγγνώμη την 185 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές. Να κάνουμε μια επαλήθευση για τη συμβαστική 8. Πως Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έμπλη 10 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 195 αποσύρθηκε. Συμβαστική τροπολογία ναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 202 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 205 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 206 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλη 3 υπέρ, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, Αποχές. Ε, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 226 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 227 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 228 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 231 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 239. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 243. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 244 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 245 αποσύρθηκε, 247 υπέρ. Κατά, αποχές, να κάνουμε μια επαλήθευση. Για την 247. Α, creo que está rechazada, pero vamos. Νομίζω ότι απερίπτεται, αλλά να το δούμε. Ρετσαθάδα. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 251 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18. Επέ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά σας παρακαλώ να... Το ξέρω ότι είναι πολλές οι ψηφοφορίες, αλλά σηκώντε το χέρι σας, γιατί αλλιώ δεν μπορώ να δω το αποτέλεσμα. Ή ε, δεν ξέρω, να το βγάζω από το μυαλό μου. Απροβάδω. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία, ε, συγγνώμη, 257 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 261 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 262 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60, 265 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έμπλη 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έμπληκος 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 34 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, άποχες, απορρίπτεται. 49 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κουλ 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Κουλ 31 ε, καλύπτεται. Κουλτ 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κουλτ 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 και 5 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 3 υπέρ κατά αποχή εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά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 Νομίζω ότι απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε τη 13. Ναι, απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, εγκρίνεται. Συγγνώμη κύριε Σεμπαστιά. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ κατά, άποχες, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 25 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, 4 αποχές. Ε, συγχαρητήρια κυρία Αρένα. Bueno, vamos a continuar. El siguiente... Συνεχίζουμε. Είναι πολύ πιο μικρή η επόμενη ψηφοφορία. Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συντάκτρια της γνωμοδότησης, η κυρία Μπιόρτερ. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 που έχει και προφορική τροπολογία που έχει ενσωματωθεί στο κείμενο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, ε, σε, δύο τμήματα, συγγνώμη, υπέρ. Α, συγγνώμη, επαλήθευση. Επαλήθευση για την 9. Rechazadas. Απορρίπτεται. 10 σε 2 τμήματα υπέρ. Κατά. Κατά, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Κατά, ε, εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές Θα κάνουμε μια επαλήθευση για τη 12. Ρετσαθάδα. Απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μία προφορική τροπολογία, την οποία... Α, συγγνώμη, δεν είναι προφορική τροπολογία, είναι αρχική παράγραφος σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές, απορρίπτεται. 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. στην 18 έχουμε και μία προσθήκη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τελικό κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. y queda aprobado por 26 votos. Εγκρίνεται 26 ψήφοι υπέρ, μία κατά και τέσσερις αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Πίερτερ. ¿Te apetece ponerte un ratito? Bueno, pues pasamos al Ωραία. Περνάμε στη γνωμοδότηση της κυρίας ε, Σταράς Φεραγκούτ για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Ξεκινούμε με την ψηφοφορία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα σουηδικά. It's okay? Yeah, okay.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 84 τέσσερα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Θέλετε να κάνουμε παλήθευση της 59. La 59 estamos rechazada. Απορρίπτεται η 59, συμβαστική τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 60 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση της 60, Δεν έχω διερμηνία. Now good. Εντάξει, εντάξει, έφτιαξε. Χωρίς μικρόφωνο, πρόεδρος. Είμαστε λοιπόν στην 60, η οποία και εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 69 ήταν ε, στον ε, συμβιβασμό 4. Έχει ενσωματωθεί εκεί. Εντάξει, συμβαστική τροπολογία 4. Και τώρα που είμαστε. Ελά, 70. Τροπολογία 70, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 με προφορική τροπολογία που έχει ε, ενσωματωθεί στο κείμενο υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές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 αποχές εγκρίνεται. 16 και 18 που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, επαλήθευση της 17, άρχεται ψηφοφορία.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το τελικό κείμενο, άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 30 ψήφοι υπέρ, μία κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Εσταράς. Pasamos a la votación de... Περνάμε στην ε, έκθεση της κυρίας Ταντσίλα για την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου στην Ευρώπη. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 4. Απροβάδο. Εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Σας παρακαλώ σηκώντε τα χέρια σας. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 και 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές ε, απορρίπτεται. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σεβαστική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το τελικό κείμενο ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Ha votado todo el Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται 17 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Νταντσίλα. Θα περάσουμε και θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση νομοδότησης όσον αφορά την πρόσθετη αξία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 αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε τον συμβιβασμό 1, συμβιβαστική τροπολογία 1. Άρχεται. Απροβάτω. Εγκρίθηκε. Και περνάμε στην τροπολογία 10, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Εγκρίνεται λοιπόν 28 ψήφοι υπέρ, 3 εναντίον. Συγχαρητήρια κυρία anche ricciute. La maratona. Περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα, που είναι η ένταξη του φύλου όσον αφορά το μηχανισμό για τη δημοκρατία. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Ολοκληρώσαμε με τις ψηφοφορίες για σήμερα. Α, Μία ανα, αναμία και όχι στο τέλο. ολικά. Σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη λοιπόν, στις 12 παρατέταρτο θα ξεκινούσε η συζήτηση με την Προεδρία του Συμβουλίου. Θα διακόψουμε λοιπόν για 15-20 λεπτά και παρακαλώ να παρακολουθήσετε στις 12 ε, παρατέταρτο στην ώρα μας ακριβώς στη συνέχιση των συζητήσεων. Vamos, vamos a reanudar con, la, con los debates. Να συνεχίσουμε με τις συζητήσεις της Επιτροπής μας. Τελείωσε η ψηφοφορία άλλωστε. Έχουμε εδώ την Προεδρία του Συμβουλίου. καλέσαμε την Ολλανδική Προεδρία από πλευρά τη Επιτροπή μα για να μα δώσει πληροφορίε σχετικά με την ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ε, Ευρωπαϊκή Στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων και τι ε, δράσει για, για τους ΛΟΑΔ. Το έγγραφο αυτό συζητήθηκε στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά δεν υπήρξε συμφωνία στο Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο ε, καλέσαμε εδώ την Προεδρία, την οποία ευχαριστούμε για την παρουσία της ε, εδώ σε αυτή τη συζήτηση. Είναι εδώ προκειμένου να μας παρουσιάσει λίγο τη συζήτηση και την παρούσα κατάσταση των θεμάτων αυτών, ώστε να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε τη συζήτηση. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο ε, Κίνγκα, εκπρόσωπο της Ολλανδικής Προεδρίας ε, του Συμβουλίου, για να κάνουμε συζήτηση μετά με τους βουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νωρίτερα, εντός του 2015, η... το Συμβούλιο Υπουργών ε, Ισότητας ζήτησε από την κυρία Γιώργα να παρουσιάσει μια στρατηγική για την ισότητα των φύλων. Το Δεκέμβριο του 2015 η Κομισιόν τελικά παρουσίασε τη νέα στρατηγική της ισότητας για το 2016-2019 με ένα έγγραφο εργασίας το οποίο ήταν η συνέχεια της στρατηγικής 2010-2015. Στη συνάντηση αυτή πολλά από τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για το καθστώς του εγγράφου εγώ και ζήτησαν μάλιστα μια ανακοίνωση και κατά την απόψή τους αυτό είναι ένα μήνυμα ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών ε, δεν είναι πλέον προτεραιότητα της Κομισιόν. Στην ε, ίδια συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου η Κομισιόν παρουσίασε τον ε, κατάλογο των δράσεων για την προώθηση της ισότητας ε, των ΛΟΑΔ. Η Κομισιόν λοιπόν εξέφρασε τις φιλοδοξίες της για τη νέα στρατηγική, για την ισότητα και για να διερευνήσει τις πιθανότητες πολιτικής στήριξης από τα κράτη-μέλη για τις ε, δράσεις αυτές ε, για τους ε, ΛΟΑΔ. Στην δήλωση της Τροϊκάς της Προεδρίας, η οποία υπεγράφει μαζί με την Σλοβεκία και την Μάλτα. Η Ολλανδία πρότεινε στα κράτη-μέλη σχέδια συμπερασμάτων του Συμβουλίου για ζητήματα φύλου και ΛΟΑΔ. Και με, τα δύο, με το να συνδυάσουμε αυτά τα ζητήματα είχαμε τρεις στόχους. Πρώτον, να επιβεβαιώσουμε την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών και για τις δύο πρωτοβουλίες της Κομισιόν. Δεύτερον, να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα για την αναγκαιότητα ένταση ε, των προσπαθειών προώθησης της ισότητας και τρίτον, να διασφαλιστεί η στήριξη όλων των κρατών μελών και στα δύο ζητήματα. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, τα περισσότερα κράτη-μέλη στήριξαν αυτή την προσέγγιση. και μπορούσαν να δεχτούν και τα δύο κείμενα ως πακέτο. Τελικά ένα κράτος μέλος είχε αντίρρηση και άρα η Προεδρία κατέληξε στο ότι δεν επετέχθη η συμφωνία. Βεβαίω η Προεδρία είναι απογοητευμένη από το αποτέλεσμα αυτό. Από την άλλη, 16 κράτη-μέλη υποστήριξαν δημοσίω ε, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για του ΛΟΑΔ, κάτι το οποίο από μόνο του είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Αναμένουμε λοιπόν να παρουσιάσουμε στο Συμβούλιο του Ιωνίου συμπεράσματα και για τα δύο ζητήματα και θα φροντίσουμε τα μηνύματα αυτά θα αντικατοπτρίζονται και τα δύο αυτά ζητήματα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Muchas Σε ευχαριστούμε πολύ κύριε Κίνγκα για αυτή την παρουσίαση. Πιστεύω ότι γνωρίζετε και έχετε συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα που από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών δίναμε και δίνουμε στη μελλοντική στρατηγική για την ισότητα των φύλων από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είχαμε μακρότατες συζητήσεις στην Ολομέλεια και την έγκριση ψηφίσματος στο Κοινοβούλιο ως προς το ότι όπως εσείς ως Προεδρία προωθήσατε στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης για να υπάρξει μεγαλύτερη πολιτική υποστήριξη και να υπάρξει μια στρατηγική ισότητα των φύλων <clears throat> και όχι μόνο η πρωτοβουλία που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ένα έγγραφο εργασίας μόνο. Για μας η σπουδαιότητα που έχει όχι μόνο είναι ο τίτλος του εγγράφου αλλά είναι είτε πρόκειται για ένα έγγραφο εργασίας είτε για μια στρατηγική. Η διαφορά είναι ότι σε σχέση με μια στρατηγική αυτή πρέπει να εγκρίνεται από το σύνολο του Κολεγίου των Επιτρόπων και γι' αυτό σημαίνει όπως εσείς το αναφέρατε μια πολιτική δέσμευση του συνόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δράσει προς αυτό το στόχο. Είμαστε και εξακολουθούμε να έχουμε συνειδητοποιήσει ότι από πλευράς των κρατών και κυβερνήσεων που υποστήριξαν αυτή την πρωτοβουλία Αναμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σημειώσει αυτή την κατάσταση και να δράσει αντίστοιχα. Σε σχέση με την, το θέμα το οποίο αντιμετωπίστηκε, σε σχέση δηλαδή με το, τα δικαιώματα συνολικά, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και έχουμε πολλές εκθέσεις με αναφορά σε αυτά πράγματι συνειδητοποιώντας ε, τι συμβαίνει με τα διαδικαστικά θέματα όσον αφορά την λήψη απόφαση από το Συμβούλιο υπάρχουν συγκεκριμένα θέματα που απαιτούν βέβαια ομοφωνία. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να προβληματιστούμε και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούν να υπάρξουν συγκεκριμένες συζητήσεις ε, που τροχοπεδούνται όμως από την θέση αυτή αποκλειστικά ενός κράτους μέλους ε, όπως ε, εσείς αναφέρατε κιόλα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μια δυνατότητα να τροποποιηθεί, να αλλάξει αυτό το θέμα αυτή η κατάσταση και να ξανααναλυφθεί πρωτοβουλία και να υπάρξει αλλαγή θέσης όσον αφορά την κυβέρνηση που σε αυτή την περίπτωση τροχοπέδησε την λήψη απόφασης. Θέλουμε όμως να σας διαβιβάσουμε το μέλημά μας, την ανησυχία μας. Ανησυχία ότι μπορούν έτσι να τροχοπεδηθούν πρωτοβουλίες που είναι σημαντικές για να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη <clears throat> που δεν πρέπει τις πολιτικές μόνο στο επίπεδο το οικονομικό αποκλειστικά να σε εξετάζει, αλλά στο πλαίσιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και όταν κάνουμε λόγο για αυτό το συλλογικό πλέγμα, κάνουμε λόγο για ένα ουσιοδέστατο θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αρχές και αξίες ε, εκείνων που θέλαμε να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση επ' αυτών της δικαιοσύνης και της ισότητας και τέτοιου είδους δράσεις αντιφάσκουν αντιβαίνουν τις ε, ουσιαστικές θεμελιώδεις αρχές στις οποίες θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτή την τοποθέτηση από πλευράς μου Προέδρου της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών ανοίγουμε τη συζήτηση Παρακαλώ θα λάβουν τον λόγο οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παρέμουν τώρα. Θα λάβει τον λόγο εξ ονόματος ε, των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα κυρία Αρετή, παρακαλώ. Oui, euh, merci, Madame euh, la Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. αντί για συγκεκριμένε ερωτήσει, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις ε, και να σχολιάσω κάποια πράγματα. Θα ήθελα να πω, το έχουμε άλλωστε πει και στο παρελθόν, ότι όσον αφορά το επίσημο καθεστώς ε, του εγγράφου το οποίο μας υπέβαλε η Επίτροπος Γιούροβα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για μια στρατηγική δέσμευση, το ΕΛΚ δεν είχε ε, κάνει ολόκληρη ιστορία για το, το τι θεωρείται αυτό το έγγραφο ε, επισήμως για τη στρατηγική, έγγραφο στρατηγικής ή όχι. Άκουσα όλα αυτά τα οποία είπαν διάφορες πολιτικές ομάδες και η Προεδρία προηγουμένως δεν ήταν και λόγος να υπερβάλλουμε και να μιλάμε συνεχώς γι' αυτό, γιατί σημασία έχει να προχωρήσουμε, να υπάρχουν συγκεκριμένε ρεαλιστικές προτάσεις και να είμαστε αποτελεσματικοί όσο μπορούμε. Και ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι η προηγούμενη στρατηγική κατά πάσα πιθανότητα δεν απέφερε όλους τους καρπούς που ελπίζαμε, ε, που προστοκούσαμε έπρεπε να προχωρήσουμε με κάπως διαφορετικό τρόπο αλλά με μεθοδικό ε, τρόπο και ρεαλιστικό τρόπο. Ακριβώς λοιπόν στο όνομα αυτού του ρεαλισμού και της ανάγκης της αποτελεσματικότητας ε, εξετάζουμε εάν υλοποιούνται ή δεν υλοποιούνται κάποια πράγματα, κυρίως για κάποια θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την πολιτική μας ομάδα και με τα οποία ε, συμφωνούμε και με άλλες πολιτικές ομάδες. Το θέμα της ε, καταπολέμησης της βίας ε, κατά των γυναικών και την πρόσβαση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. συμφωνούμε με όλα όσα γίνονται προκειμένου να προσχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και να την υπογράψει και πρέπει όλα τα θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν το αμφισβητούμε αυτό, υποστηρίζουν αυτό το ε, σημείο πρόοδου το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θεωρούμε ότι θα ε, είναι και μεταδοτικό για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμα δεν έχουν υπογράψει και κυρώσει και θέσει και σε εφαρμογή ε, για αυτούς που έχουν κυρώσει και υπογράψει όλες τις δεσμεύσεις της Σύνθηκης της Κωνσταντινούπολης. Θεωρούμε ότι εκεί έχει υπάρξει κάποια πρόοδος και γι' αυτό ε, υπεύθυνα είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το σχέδιο οδηγίας λέει ε, Women on Boards, ε, ε, γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Εμείς ως ΕΛΚ δεν είμαστε η μόνη πολιτική ομάδα που έχουμε στεναχωρηθεί για αυτή την στασιμότητα που υπάρχει και το γεγονός ότι έχει μπλοκάρει η υπόθεση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Για μας ε, είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί ε, πλέον και κάτι το οποίο έχει προσλάβει συμβολικό χαρακτήρα για να μπορέσουμε να ε, δίνουμε μεγαλύτερες ευθύνες ε, στις γυναίκες ε, σε διευθυντικές θέσεις. Και ένα άλλο θέμα για το οποίο το ΕΛΚ ανησυχεί πολύ και ταυτόχρονα παρακολουθεί και τι μπορεί να υπάρξει, αν υπάρχουν νέες προτάσεις, νέοι δρόμοι υπάρχει το θέμα του gender pay gap, ε, της διαφοράς μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών ε, και προσπαθούμε να κάνουμε την κατάλληλη διάγνωση για να δούμε τι ανισότητες υπάρχουν και στα ε, συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών και να προτείνουμε και συγκεκριμένα μέτρα και ρεαλιστικά μέτρα. Αυτά λοιπόν για την ε, πολιτική μου ομάδα είναι ήδη παρατηρήσεων και ε, θα πάρουν το μέρος και άλλες μέλη της ομάδας. Σας ευχαριστούμε. Εξ ονόματος της ομάδας η κυρία Θετσέρα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Προσυπογράφω πλήρως πρόεδρε τα σχόλια που έγιναν από πλευρά της Προεδρίας. Έχουμε μια συμφωνία που είναι πάρα πολύ σημαντική, κέρια σημασία όσον αφορά την ισότητα, τα θέματα ισότητας θεμελιώδες δίκαιο όσον αφορά τη δράση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω ρητά εξ ονόματος φιλελεύθερης ομάδας για τα όσα έγιναν και αναφέρθηκαν από την Ολλανδική Προεδρία σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Έχοντας πετύχει ότι 27 από τα 28 κράτη-μέλη συμφωνούν τουλάχιστον σε αυτή την κοινή προσπάθεια προσέγγισης είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτό. Θέλω επίσης όμως να τονίσω ότι κάνουμε λόγο για την Ουγγαρία κράτος μέλος που, που τροχοπέδησε και απέριψε λόγω αυτής της απόρριψης την λήψη αυτής της απόφασης. Είναι η Ουγγαρία λοιπόν, μια χώρα που με συνέπεια διαρκώς σε σχέση με αυτές τις ε, καταστάσεις ε, δραστηριοποιείται Δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει όμως να σέβεται τις ε, δεσμεύσεις που έχει ένα κράτος όταν επιθυμεί να ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν οι επιφυλάξεις της Ουγγαρίας ότι δεν είναι σε θέση να συμφωνήσει με τον κατάλογο δράσεων σε σχέση με τα θέματα αυτά ε, θα πρέπει πολύ σοβαρά να το πάρουμε υπόψη αυτό το ζήτημα εμείς αυτές τις δράσεις δηλαδή που η Επιτροπή είχε προτείνει ως στόχο το Δεκέμβριο του 2015 <clears throat> με τις ε, με προοπτικές ε, το 2017-2019 όλα αυτά συνέβησαν μετά από την ε, διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπό το φως των στοιχείων που είχαν συλλεγεί όσον αφορά τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων Πρόκειται για μια δέσμευση λοιπόν και για ένα κατάλογο δράσεων που δεν είναι κατά το δοκούν συντάχθηκε, είναι συνενετικά προσεγγίστηκε και ε, συντάχθηκε. Και αναμένουμε το 2008 να εξετάσει το Συμβούλιο την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία για την ισότητα αντιμετώπισης των φύλων και αληθεύει ότι αυτή η οδηγία επίσης ε, προέβλεπε και τα θέματα διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά τα θέματα υπηρεσιών για παράδειγμα να μην υπάρχει καμία αρνητική διακριτική μεταχείριση λόγω θρησκείας ειδικών αναγκών ατόμων με ειδικές ανάγκες κοινωνικής κατάστασης, κοινωνικής κατάστασης και υγείας όσον αφορά την εκπαίδευση, την παιδεία και την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και στη ακόμα. Και πάλι αληθεύει εδώ ότι υπάρχει μια πτυχή που δεν ε, συμπεριλαμβάνεται σε σχέση με τις δράσεις κατά της ε, αρνητικής μεταχείρισης ε, για τους διεμφυλικούς, για παράδειγμα. Αλλά θα θέλαμε να εμείνουμε για τη σπουδαιότητα που έχει, κυρίως σε ένα πλαίσιο που έχει κέρια σημασία, όπως η ισότητα, που πρέπει οπωσδήποτε το παλαιό άρθρο 2 3 της ε, Χάρτας ε, των Δικαιωμάτων για την ισότητα συνολικά να, ε, να εφαρμόζεται. Αυτή η απουσία συμφωνίας οφείλεται στην απόρριψη μιας χώρας που συστηματικά με συνέπεια δείχνει ότι δεν συμφωνεί να δεσμεύεται από τα συμφωνημένα, συμπεφωνημένα και βλέπουμε λοιπόν αυτό το ότι έχει αυτό τον ξεχωριστό χαρακτήρα. Από την άλλη πλευρά, σε σχέση με την οδηγία για τις γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, θα ήθελα να αναφέρω ότι πήρα μία απάντηση σε μία ερώτηση που είχε κατατεθεί από πλευράς του Συμβουλίου, από αυτή την Προεδρία του Συμβουλίου, στην οποία απάντηση αναφέρεται ότι η Ολλανδική Προεδρία αναλύει πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από νομικής, νομοθετικής πλευράς αυτό το θέμα για να μπορέσει να προαχθεί <clears throat> όταν και εφόσον υπάρχουν ε, ενδείξεις για, για μια αλλαγή της κατάστασης και των όρων από το 2015. Θα θέλαμε εδώ να υπάρξει αυτή η αναφορά σε ποιες πτυχές ε, και σε σχέση με τον αριθμό των χωρών, ε, σε σχέση με την απόρριψη προτάσεων, αν υπήρξε πρόοδος ή όχι και ποιες προοπτικές και ποια σημασία έχει όλο αυτό διότι σε σχέση με το έργο της προαγωγής αυτής της οδηγίας ακριβώς είχαμε το θέμα της Ολλανδίας ε, που είχε κέριο ε, ρόλο και επί, στο τέλος να αναφέρω ότι υπάρχει μια πτυχή που είναι σημαντική σε σχέση με την Προεδρία και εσείς ε, το τονίσατε αυτό επίσης για τη συνέχεια που πρέπει να υπάρξει για αυτό το έργο από τις επόμενες Προεδρίες αυτή η συνέχεια που πρέπει να διασφαλιστεί είναι κέρια σημασία. Ξεκινάμε με βάση ένα σημαντικό έργο που έχει επιτελεστεί κατά το παρελθόν και πρέπει να διασφαλιστεί η συνέχειά του. Και στον καθορισμό των θεμάτων είναι σημαντική οι όροι, οι, τα, με, οι διατυπώσεις, οι όροι περιγράφουν αυτά τα πλαίσια και γι' αυτό η, η πλειοψηφία ε, για την ευρωπαϊκή στρατηγική πρέπει να ε, προχωρήσει με βάση αυτές τις αρχές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπεθέρα. Η κυρία Μπιόρκ παρακαλώ για την ενωτική αριστερά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο διάλογος και σημαντικό για το Συμβούλιο και την Προεδρία να ε, έχουν αυτή την ευθύνη να έρθουν εδώ και να μας ε, συναντήσουν. Έχετε δίκιο, υπάρχει αυτή η δήλωση του τρίου της ε, Προεδρίας, αλλά βλέπουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέτωπο της ισότητας. Οι γυναίκες το βλέπουν, βλέπουν ότι υπάρχει καταστροφή. Δεν γίνεται τίποτα για την ε, γονική άδεια ή την άδεια μητρότητας. Εμείς στη Σουηδία ε, δεν βλέπουμε καμία σοβαρή αλλαγή. Κάποια πράγματα θα μπορούσαν να είναι τόσο θετικά για τις γυναίκες, ε, αλλά κολλάνε όλοι στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Καλοδεχούμενη λοιπόν η δήλωση της Προεδρίας και η προσπάθεια που κάνατε δεν είμαστε πολύ ικανοποιητικοί ή ικανοποιημένοι με για το ότι η Ουγγαρία κατάφερε να μπλοκάρει ε, από μόνη της τα συμπεράσματα. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να υπάρξει κάποια λύση των Ιούνιο θα καταπολεμήσετε αυτές τις ε, μη φιλικές προς τις γυναίκες απόψεις στο Συμβούλιο. Και βεβαίως ε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ ενός εγγράφου εργασίας ε, εσωτερικού και ενός εγγράφου στρατηγικής. Νομίζουμε πως με αυτά συμφωνούν όλοι και εκτός του Κοινοβουλίου η Κομισιόν επιδεικνύει αλαζονία με το να μην φέρνει αυτό το έγγραφο το οποίο ζητάει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Κάθονται εκεί στην Κομισιόν και λένε όχι. Δεν θα ασχοληθούμε με τέτοια πράγματα. Απαράδεκτο. Θα δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Για να προχωρήσει η κατάσταση πρέπει κάτι να γίνει εδώ. Ευχαριστώ κυρία Μπιόρκ. Εξ ονόματος των Πρασίνων, η κυρία Ρέπκε, παρακαλώ. Uh, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ από πλευρά μου, λέει η κυρία Ράνικε, για αυτό το διάλογο. Για να είμαι ειλικρινής, θα πήγαινα πιο πέρα από τη συνάδελφο της Γκουε, της Ενωτικής Αριστεράς όχι μόνο σε σχέση με μια τοποθέτηση, αλλά βλέπουμε και μια οπισθοδρόμηση ένα πισωγύρισμα σε σχέση με τα θέματα της ισότητας και την οριζόντια οδηγία, την ε, οδηγία για τη μητρότητα και την γονεϊκή άδεια. Όχι μόνο δεν προχωράμε, αλλά έχουμε και μια οργανωμένη, ενορχιστρωμένη επίθεση κατά των δικαιωμάτων των γυναικών και απογοητεύομαι με την αντίδραση που έχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για αυτή την επίθεση που έχουμε υποστεί. Και είχα και τις ελπίδες ότι όταν ε, ξεκίνησε αυτή η Επιτροπή κατά την έναρξη της Προεδρίας ότι θα σημειώναμε πρόοδο, αν όχι σχέση με τα ε, θέματα της ισότητας, οδηγίας για την ισότητα, για τα θέματα αυτά, τα συγκεκριμένα τώρα. Και τώρα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου η άλλη πλευρά θα έλεγα, η άλλη όχθη, Μόνο ένα κράτος μέλος έχει τροχοπεδίσει οποιαδήποτε κίνηση και κινητοποίηση. Και τι κάνουμε, έχουμε μόνο συμπεράσματα προεδρίας. Επαρκεί αυτό. Όχι, πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι η στρατηγική για να αντιστραφούν οι όροι αυτής της κατάστασης, αυτού του παιχνιδιού ποιες προσπάθειες μπορούν να αναλυθούν για να καταλήξουμε σε μια επίλυση αυτού του πολύ σημαντικού προβλήματος. Γιατί έχουμε μια προεδρία πάλι, πάλι οπισθοχωρούμε, υπαναχωρούμε και όχι μόνο δεν θα σημειώσουμε πρόοδο, αλλά θα εγκαταλείψουμε, θα απεμπολίσουμε πολύ σημαντικά θέματα και δικαιώματα του ανθρώπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαράδεκτο αυτό. Θα ήθελα από την Ολλανδική Προεδρία να δούμε τι μπορεί να γίνει και πώς μπορούμε εμείς να δράσουμε, να αλλάξουν τα πράγματα, να βρισκόμαστε τον Ιούνιο πάλι εδώ και ακούσουμε ότι μόνο τα συμπεράσματα της Προεδρίας είναι εκείνα περί των οποίων πρόκειται. Απεμπολούμε δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά είναι απόλυτα αναγκαίο. Ίσως θα μπορούσαμε να ακούσουμε περισσότερο ποιες ιδέες έχετε και υπάρχουν, ώστε εμείς σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή που στεναρότατα υποστηρίζουμε την ισότητα των φύλων, να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ρέτκε. Και για να ολοκληρώσουμε έχετε εσεί τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστώ και το Συμβούλιο <clears throat> λέει η κυρία Μπεθερίλ και για το Συμβούλιο ευχαριστώ για αυτό το διάλογο με την Επιτροπή μας. Και εξίσου όπως όλες οι συνάδελφοι και η συντονίστρια της ε, ομάδας ε, που παρενέβη προηγούμενα αναφέρθηκαν τα πιο σημαντικά θέματα όπως για παράδειγμα την έγκριση της ε, συμφωνίας της Κωνσταντινούπολης και σε αυτή την ομάδα για την καταπολέμηση της ε, βίας ε, με βάση το φύλλο και προωθούμε ως προτεραιότητα ως Κοινοβούλιο αυτό που έχουμε ως προτεραιότητα όλοι οι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο και το θέμα των μισθολογικών διαφορών, του μισθολογικού χάσματος εις βάρος των γυναικών αυτή τη φορά και να δούμε και την ανάδειξη γυναικών σε θέσεις ε, που θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις όπως τα διοικητικά συμβούλια Women on Board. Και μια άλλη οδηγία που έχει τροχοπεδηθεί για την ε, οδηγία για τη μητρότητα κάνω λόγο. Και ένα άλλο θέμα το οποίο μας ανησυχεί και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αλλά επίσης ε, αυτό με το οποίο ασχολούμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή με τα θέματα των θυμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω την Ολλανδική Προεδρία για το ότι μία από τις προτεραιότητες της πραγματική προτεραιότητα είναι η υποστήριξη των θυμάτων, κάθε είδους θυμάτων, όλων αυτών των εγκλημάτων και παραπτωμάτων και από πλευράς της Ολλανδικής Προεδρίας ακριβώς με κάθε τρόπο η υποστήριξη των δικαιωμάτων των θυμάτων. Μια και ήμουν εισηγήτρια και τώρα υλοποιούμε τα θέματα της οδηγίας για την υποστήριξη, προστασία και ενδυνάμωση των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων είναι πολύ σημαντικό ως ε, Επιτροπή Γυναικών μέσα στο πακέτο μέτρων κατά της βίας εις βάρος των γυναικών να δράσουμε. Είναι πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση που έχει αναπτύξει το Συμβούλιο για αυτά τα θέματα ώστε να μπορέσει αυτή η οδηγία και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Εντολή για την προστασία των θυμάτων να προχωρήσουμε για την υλοποίηση ακριβώς και εφαρμογή όλων αυτών των θεμάτων στην πράξη τώρα. Και θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε όλα αυτά όλα όσα αφορούν την, το λαθρεμπόριο ανθρώπων, το εμπόριο ανθρώπων και συντριπτική πλειοψηφία αυτών των θυμάτων ανθρωποεμπορίας είναι γυναίκες και παιδιά για σεξουαλική εκμετάλλευση θύματα δηλαδή πάλι. Είχαμε και την έκθεση για την εφαρμογή αυτής της ε, οδηγίας ε, και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να τα δούμε αυτά. Θα ήθελα να έχουμε περισσότερες αποσαφηνήσεις, επεξηγήσεις για τα θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Θέματα ταμπού, ακόμα και τα θέματα πορνείας για παράδειγμα με βάση τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά και όλα όσα συσχετίζονται σε σχέση με τα σεξουαλικά θέματα και την προστασία των γυναικών και των θυμάτων. Να ε, καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες και να είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των θυμάτων του ανθρωποεμπορίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπεθερίλ. Και μετά από αυτή την ε, τον γύρο σκέψεων και παρατηρήσεων που έγινε από τις ε, βουλευτίνες ε, ο κύριος Κίνγκα θα λάβει τον λόγο για να απαντήσει πιο εξειδικευμένα στις παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνούμε με τις ανησυχίες σας για το ότι κάποιες διαδικασίες εντός του Συμβουλίου ε, είναι τροχοπέδι στην πρόοδο για τις παρατηρήσεις του ΕΛΚ. Οπωσδήποτε συμφωνούμε ότι ανεξαρτήτως ε, της ε, φύσης των διαφόρων ανακοινώσεων ή εγγράφων μας έχει η πρακτική πρόοδος. Για την βία κατά των γυναικών ε, μας απασχολεί πάρα πολύ και εργαζόμαστε σκληρά. Επίσης ε, τα ζητήματα για τις γυναίκες στα ΔΣ ε, για το ΕΛΚ ε, και τους φιλελευθερούς. Κοίταξε, ας είμαστε σαφείς. Εμείς είμαστε διαμεσολαβητές εδώ πέρα. Και μόλις λάβουμε κάποιο μήνυμα τα πράγματα αλλάζουν στα κράτη-μέλη θα το προχωρήσουμε. Αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμα τέτοιο μήνυμα. Γιατί όπως σας είπα εμείς μεσολαβητές είμαστε. Γι' αυτό ακριβώς ε, δεν έχουμε προχωρήσει. Μετά για το θέμα του χάσματος ε, στις αμοιβέ και στις συντάξεις είναι οπωσδήποτε ένα κομμάτι του εξαμήνου πλέον και άρα επαφιέται στα κράτη-μέλη να κάνουν τα δέοντα. Για τις άλλες παρατηρήσεις ε, της Άλντε σας ευχαριστώ για την στήριξή σας. Για το θέμα της ισότητας ε, πέρα από τον τομέα της εργασίας προσπαθήσαμε να προωθήσουμε το ζήτημα και για τη συνεργασία με τη Σλοβακία και τη Μάλτα ε, υπάρχουν οι δηλώσεις ε, της Τρόικας της Προεδρίας και βεβαίως ε, θα φροντίσουμε τα όσα κάνουμε εμείς στη δική μας Προεδρία να συνεχιστούν και στις επόμενες. Μετά, η βουλευτής ε, της ΓΚΟΕ ε, ρώτησε για το θέμα της γονικής άδειας, της άδειας πατρότητας. η Κομισιόν ετοιμάζει τις προτάσεις της, νομίζω θα είναι έτοιμες μέχρι το τέλος του έτους. Βεβαίως, υπήρχαν πολλές ερωτήσεις για τις προθέσεις ε, της ε, Προεδρίας ε, σε σχέση με τα συμπεράσματα για τους ΛΑΡ και την ισότητα. Βεβαίως, Είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Από την πρώτη μέρα όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν ότι όλα αυτά πρέπει να είναι πακέτο. Όπως είπα, προετοιμάζουμε συμπεράσματα της Προεδρίας για το Συμβούλιο του Ιουνίου, αλλά συμφωνούμε μαζί σας ότι καλό είναι να έχουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου και είμαστε και σε στενή επαφή με τα υψηλότερα πολιτικά επίπεδα στα κράτη-μέλη για να δούμε εάν ε, μπορούμε να διορθώσουμε την κατάσταση και να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που ήταν η αρχική μας ε, πρόθεση. Είναι θετικό το ότι το στηρίζετε και ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε εγώ θα έλεγα προσπαθήστε να επηρεάσετε την κυβέρνησή σας. Και οι πράσινοι το έφτιαξαν. Γενικά σας ευχαριστώ για την στήριξή σας για να το έχουμε ένα πακέτο το ζήτημα. Και σας ευχαριστώ και για τις ε, παρατηρήσεις σας και τις ερωτήσεις σας που δείχνουν το πόσο σοβαρά παίρνετε το θέμα. Και έλαβα το μήνυμα της στήριξης ε, προς την Προεδρία και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτονόητο Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ ανάμεσά μας για αυτή τη συζήτηση και χωρίς αμφιβολία θα δούμε με ποιες δράσεις από την Επιτροπή μας μπορούμε να προχωρήσουμε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε στο τέλος μια αποτροχοπαίδηση, μια απελευθέρωση αυτού του θέματος όσον αφορά τα δικαιώματα ε, κυκλοφορίας ε, και δράσεις. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πολλές φορές ο χώρος για να ελιχθεί αυτό το Ευρωκοινοβούλιο για ελιγμούς είναι πολύ περιορισμένος. Αλλά τουλάχιστον ότι υπάρχει μια πολιτική εδώ τοποθέτηση είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθεί αυτή η πρωτοβουλία από πλευρά της Προεδρίας. Θα δούμε ποιες δυνατότητες υπάρχουν για κάποια ανάληψη δράσης προηγούμενα ώστε να μπορέσετε εσείς σε σχέση με το Συμβούλιο να δώσετε συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε διακόπτουμε τη συνεδρίασή μας. Θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα <clears throat> με την κυρία Ζούροβα από πλευράς Επιτροπής μας. Γεια σας.